Thank you. We start immediately. Λοιπόν, συνεχίζουμε αμέσως με το επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη, που είναι ε, θέματα ασφαλείας, πτυχές σχετικές με την ασφάλεια στις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Ασίας. Η κυρία Σουίτσα. Έχουμε το σημείο 5 τώρα. Πού είναι οι σχέσεις μας με την ε, Κίνα για το θέμα αυτό. Κύριος Στίβεν Εβερτς που είναι επικεφαλής σύμβουλος και κυρία Πάισοβα που είναι επικεφαλής αναλήτρια από το Ίδρυμα για τις ε, Μελέτες Ασφάλειας. Να ξεκινήσω λοιπόν με μια εισαγωγή και να σας πω πως αυτή η κοινή συνάντηση ξεκινά μια πολύ επίκαιρη συζήτηση για το πώς θα εξελιχθούν περαιτέρω οι στρατηγικές Ευρωπαϊκής Ένωσης, να έχουμε μεγαλύτερη συμμετοχή και μεγαλύτερη παρουσία ε, στο θέμα της ασφάλειας και της ειρήνευσης στη Νότια και στη Νοτιοανατολική Ασία. Είναι σημαντικό και για την παγκόσμια ειρήνη και την παγκόσμια ασφάλεια και αυτό αναγνωρίζεται στα πλαίσια της στρατηγικής ε, της ε, Ευρώπης. Χρειάζεται περισσότερη συνεργασία με την Ασία, ε, θαλάσσιες μεταφορές, άλλες μεταφορές, κυβερνη, κυβερνοασφάλεια, ειρηνευτικές αποστολές, αντιτρομοκρατία, μάχη κατά του εξτρεμισμού και μάχη για την αποφυγή της διάδοσης των πυρηνικών, βιολογικών και χημικών όπλων. Μην ξεχνάτε ποιες είναι οι παγκόσμιες απειλές για την ασφάλεια είναι η ασφαλεία της ενέργειας, είναι το καθαρό νερό, είναι οι πανδημίες, είναι ε, το κλίμα. Το 2018 το Συμβούλιο υπέγραψε τα συμπεράσματα για την ε, ενισχυμένη συνεργασία με την Ασία για να εξασφαλίσουμε ε, συστήματα που θα βασίζει το κράτος δικαίου, πολυμερή συστήματα, περιφερειακή σταθερότητα, δικαιώματα των πολιτών μας και βεβαίως να εξασφαλίσουμε τα ευρωπαϊκά οικονομικά συμφέροντα. Οι ευρωπαϊκοί θεσμοί και τα κράτη-μέλη συντονίζονται περισσότερο και είναι ε, πιο συντονισμένοι με τους ασιατικούς, ε, με τους εταίρους από την Ασία, έτσι ώστε να έχουμε οικοδομήσει δυναμικού στη σχέση μας με την Αζιάν και την Ασία. Η συμμετοχή στα φόρουμ αυτά, τα περιφερειακά, είναι ε, κομβικά για τα συμφέροντά μας πέρσι, για την ελευθερία της πλοήσης στην θάλασσα της Νότιας Κίνας και για την μη αναγνώριση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κίνας, στα πλαίσια αυτά ε, έπλεσαν ε, ε, ο Αγγλικός και ο Γαλλικός στόλος στα ύδατα τα οποία διεκδικεί η Κίνα. Το ίδιο έχουν κάνει και οι Ιάπωνες και οι Αμερικάνοι. Δεδομένης της στρατηγικής σημασίας της ε, αυτή τη διαδρομή θα πρέπει να προωθήσουμε περισσότερο μια ειρηνευτική επίλυση αυτής της διαφοράς σεβόμενη πάντα το διεθνέ δίκαιο. Για το ρόλο της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης στις ε, συνομιλίε Βορείου και Νοτίας Κορέα, δεν νομίζω ότι περιμένει κανεί, εμεί να έχουμε λύση, να έχουμε θέση διαιτητή, αλλά μπορούμε τουλάχιστον να διευκολύνουμε αυτέ τι συνομιλίε. υπαρχουν Υπάρχουν αρκετά ευρωπαϊκά κράτη-μέλη τα οποία έχουν στην Pyongyang πρεσβείε και μπορούν να μεταφέρουν μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών μηνύματα. Μπορούμε επίση να προσφέρουμε τον τόπο για συναντήσει υψηλού επίπεδου, αλλά θα πρέπει να συνεχίσουμε μια στεναρή πολιτική κυρώσεων μέχρι να έχουμε απτά ε, αποτελέσματα, επαληθεύσιμα αποτελέσματα στην αποπυρηνικοποίηση της ε, Βορείου Κορέας και αν δούμε θετικά αποτελέσματα θα πρέπει εμείς να στηρίξουμε την εφαρμογή των συμφωνιών και να έχουμε ε, και να προσφέρουμε ανθρωπιστική βοήθεια σε μια επόμενη φάση. Αυτά ως εισαγωγή. Τώρα θέλω να ξεκινήσουμε με την ανταλλαγή απόψεων. Κυρία ε, Φωτίγκα, μπορείτε να καλωσορίσετε ε, τους προσκεκλημένους μας. Βεβαίως. Άφετ και Σέντε λοιπόν συνεδριάζουμε από κοινού μαζί. Είδατε ε, τα όσα μας είπε η κυρία Σουίτσα που έχει τη συμπροεδρία. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να σας παρουσιάσω τους αξιότιμους προσκεκλημένους. Είναι ο επικεφαλής ε, σύμβουλος στη συνάντηση Ασίας Ευρώπης στα πλαίσια της Υπηρεσίας Εξωτερικής Πολιτικής ο κύριος Στίβεν Έβερτς και έχουμε επίσης και την δόκτορα Εύα Πέισοβα που είναι πολύ γνωστή σε εσά. Νομίζω ήσασταν παρούσα δύο, σε δύο ή τρεις συναντήσεις της ΕΔΕ και ακούσαμε πραγματικά άριστες παρουσιάσεις από πλευρά σας για τις προκλήσεις που δημιουργούν κυρίως η Κίνα αλλά και άλλοι στην νοτιοανατολική Ασία και τα πλαίσια της, ε, ε, των όσων συμβαίνουν στην ε, θάλασσα της Νοτιοκίνας. Σας, καλούμε, σας ε, καλωσορίζουμε εδώ, είστε επικεφαλής αναλήτρια και σας ε, καλωσορίσουμε στο πάνελ και στη συζήτηση. Χωρίς λοιπόν να καθυστερώ τη συζήτηση, κύριε Στίβεν Εύερτς έχετε το λόγο. Εδώ βλέπω να μην έχετε αλλάξει τη σειρά μεταξύ σας. Ό,τι επιθυμείτε, κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Είμαι πολύ ικανοποιημένο που έχουμε αυτή την ευκαιρία να κάνουμε μια ανταλλαγή απόψεων για τη στρατιωτική ε, δέσμευση που έχουμε αναλάβει στην ε, Νότιο-Ανατολική Ασία είναι κάτι καινούριο, θα είμαστε ειλικρινεί, αλλά αναπτύσσεται συνέχεια και είναι καλό που θα κάνουμε την ανταλλαγή απόψεων για να δούμε τι έχει συμβεί ήδη και τι έπεται. Να σας υπενθυμίσω λοιπόν, για να ε, βρισκόμαστε όλοι στο ίδιο, στην ίδια φετηρία, γιατί και για ποιο λόγο αυξημένη ε, συνεργασία με τους εταίρους μας στην Νοτιοανατολική Ασία. Ξεκινήσαμε από το γεγονό της αναγνώρισης πως έχουμε ε, όλοι συμφέροντα από την ασφάλεια του άλλου. Ζούμε σε ένα περιβάλλον παγκοσμίου ασφάλειας, ό,τι συμβαίνει και επηρεάζει εμά και αντίστροφα. Επίσης, ασφάλεια και οικονομία γιατί οι συζητήσεις με την Ασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνήθω ξεκινάνε με τις εμπορικές οικονομικέ σχέσεις που είναι πολύ σημαντικέ για μα, Επενδύσεις όμως και εμπόριο με την Ασία, όλα αυτά βασίζονται στο γεγονός που θα έχουμε συνεχιζόμενη στρατηγική σταθερότητα στην περιοχή. Οπότε υπάρχει αυτή η σύνδεση μεταξύ οικονομία οικονομίας και ασφάλεια. Ε, στις σχέσεις που διέπουν την Ευρωπαϊκή Ένωση με την Ασία. Είναι ένας κόσμος ο οποίος αλλάζει συνέχεια, μεταλλάζεται με κάποιες πιο βαθιές τάσεις επειδή έχουμε κάποιες αλλαγές ε, στα όσα συμβαίνουν εκεί στην περιοχή και βέβαια στην κορυφή έχουμε τις ταχύτητες εξελίξεις που έχουν να κάνουν με το ρόλο των ΗΠΑ και που επηρεάζουν και αυτές τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλα αυτά λοιπόν αιτιολογούν το γιατί γίνεται μια όλο και περισσότερη και βαθύτερη συζήτηση και υπάρχει ε, και το σχετικό αίτημα των εταίρων μου στην Ασία να έχουμε πιο δραστήρια δράση. Βέβαια, ο δικός μας ρόλος είναι πολύ διαφορετικός από αυτόν τον είπα ή άλλων μεγάλων παικτών, αλλά νομίζω στα μάτια τους έχουμε μία προστιθέμενη αξία ακριβώς γιατί οι άλλοι παίκτες έχουν πολύ πιο ισχυρά πολιτικά, ε, στρατιωτικά προφίλ. Ε, εμείς έχουμε τα δικά μας συμφέροντα, το δικό μας, τη δική μας ταυτότητα στα θέματα ασφάλειας ε, και πολιτικής και γι' αυτό είναι και ευδιάκριτος ο ρόλος μας. Και επειδή αναφερθήκατε στα συμπεράσματα του Συμβουλίου προηγουμένω, είπαμε ενισχυμένη συμμετοχή στα θέματα ασφάλειας στην και με την ε, Ασία. Ε, δεν πρόκειται για τυπογραφικό λάθος. Έχουμε μεγαλύτερη συμμετοχή στην Ασία, ναι, αυτό είναι σημαντικό, αλλά μαζί με τους Ασιάτες εταίρους μας. Εμείς εκεί, αλλά όχι μόνο εκεί, στο χώρο ε, μεταξύ μας και στην παγκόσμια σκηνή. Δεν ξεκινάμε από το τίποτα. Τα τελευταία χρόνια έχουν συμβεί πολλά και έχουμε ενισχύσει σε μεγάλο βαθμό τη συνεργασία μας και θα αναφερθώ ε, στα όσα κάναμε στο ΑΤΣΕ πριν από χρόνια, ειρηνευτικέ αποστολέ και ο, ο τρόπο με τον οποίο λειτουργούν σε όλη την περιφέρεια. Και αυτό είναι σημαντικό αν δείτε τι κάναμε και στο Μιντανάο, στη Μιανμάρ, με την Κίνα Έχουμε ένα συνεχιζόμενο διάλογο ε, για την ασφάλεια σε πολλά επίπεδα. Η ΥΠΑΤΗ εκπρόσωπος, η Υπουργό Άμυνας και βεβαίως και την κλιμακωτή ε, συζήτηση που αναγνωρίζει και τα συμφέροντά μας αλλά και τους περιορισμούς που υπάρχουν. Η Ιαπωνία. Βλέπουμε πώς μπορούμε ε, ε να συνεισφέρει ε, τουλάχιστον ε, στις ειρηνευτικές αποστολές ε, στις, με στρατεύματα ή η Ιαπωνία στα πλαίσια της κοινή πολιτικής άμυνας και ασφάλειας. Θα γίνει αυτό το μήνα μία συνάντηση. Έχουμε το πλαίσιο Συνεργασία στρατιωτική με την Κορέα, έστειλε στην Ανταλάντα ε, ε, στόλο. Επίσης, ε, στην Ινδία, οι ειρηνευτικέ αποστολές τρόφιμα. Πακιστάν επιθυμεί να συνεργαστεί μαζί μας στο ευρύτερο πλαίσιο της επιχείρηση Αταλάντα η ΑΣΕΑΝ είναι σημαντικός σύμμαχος, κομβικός για την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί μιλά για διεθνούς κανόνες, διαβούλευση, ε, πρόσβαση για όλους, πολυμερείς συζητήσεις και ε, έχουμε ενισχύσει ε, τη συνεργασία μας στην αντιτρομοκρατία, στις επιχειρήσεις διάσωσης και στηρίζουμε και τις δικές τους προσπάθειες σε τέτοιου είδου επιχειρήσει. Θαλάσσια ασφάλεια. Εύα Πέσοβα, είστε εδώ σήμερα και χαίρομαι πολύ και κυρίως, όχι μόνο γι' αυτό βέβαια, αλλά γιατί ήσασταν εκεί από την αρχή ε, στην προσπάθεια να ενισχύσουμε τη σχέση με την ΑΖΕΑΝ για τις θαλάσσιες, την ασφάλεια στις θαλάσσιες μεταφορές, διάλογος από το 2013 σε τακτά χρονικά διαστήματα για την ανταλλαγή διδαγμάτων από περιφερειακή σκοπιά για τα συστήματα παρακολούθησης, για το IUU και για την ανάπτυξη δυναμικού στο Περιφερειακό Φόρουμ της ΑΣΕΑΝ. Εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε την συμπροεδρία με το Βιετνάμ και, το και την Αυστραλία, το σκέλος για τη θαλάσσια, την ασφάλεια θαλάσσιες μεταφορές μέχρι το 2020 και με την ΑΣΕΑΝ και μέσω του ε, Ευρωπαϊκού Στρατιωτικού και ε, Κολεγίου και Κολεγίου Άμυνας έχουμε ε, προσπαθήσει να τους εξηγήσουμε πώς λειτουργεί αυτό και να μεταφέρουμε στους εταίρους της ΑΣΕΑΝ το εξή μήνυμα. Μπορεί κανείς να οργανώνει με σοβαρό τρόπο συνεργασία, ασφάλεια και άμυνα περιφερειακό επίπεδο χωρίς να χρειάζεται να περάσεις μέσω ε, της ψηφοφορίας με ε, πλειοψηφία, γιατί δεν το επιθυμούν. Και ε, αυτό λόγω των πιέσεων που αντιμετωπίζουν πολλές φορές από ΙΠΑ, <coughs> Ιαπωνία και Ρωσία. Άντε είναι μια περιφερειακή, ένα περιφερειακό φόρουμ που αναπτύσσεται, έχουμε πει πως θέλουμε να συνεισφέρουμε και να είμαστε ένας εταίρος με θετικό πρόσημο εν ευθέτω χρόνο και στα πλαίσια αυτά θα συνεισφέρουμε και στο EDM SYN ως παρατηρητές στις διάφορες ομάδες εργασίας ε, για να εξεδιπλώσουμε τη στρατηγική μας εταιρική σχέση με τις χώρες του ΑΣΕΑΝ που αποτελεί και τον απότερο πολιτικό στόχο. Στα πλέσματα στα πλαίσια του συμπεράσματος των, ε, του Συμβουλίου Γενικών Πολιτικών Επιθέσεων ξέρετε πως έχουμε και τις σχέσεις ε, people to people, από λαό σε λαό. Ο στρατηγός Κωνσταράκος που ήταν ε, επικεφαλής στο παρελθόν ταξίδευσε πάρα πολύ για να ανοίξει αυτό το διάλογο με τα στρατιωτικά ε, με τους στρατιωτικούς κύκλους στην Ασία, όπως και με ε, υπόλοιπους, ε, με, όπως έχουμε ανοίξει και, άλλες, και άλλους διάβλους διαλόγου, η συνεργασία σε αυτό το επίπεδο είναι πάρα πολύ σημαντική. Μαρ και άλλοι εταίροι, το μήνυμα είναι πως θα πρέπει τα στρατιωτικά σώματα να ελέγχονται από πολιτικό προσωπικό και ο στρατηγός κ. Κωσταράκος και προσωπικά και εκπροσώποντας την Ευρωπαϊκή Ένωση είχε πολύ σημαντικό ρόλο που, ανάλαβε, που, που είχε αναλάβει πέρσι μας επισκέφτηκε και ο επικεφαλής ε, του Γενικού Επιτελείου Στρατού από το Βιετνάμ. Είναι σημαντικό να συμμετέχει το Βιετνάμ σε αυτά τα συμφωνίες πλαίσιο γιατί ανοίγει δρόμους για μεγαλύτερη επιχειρησιακή συνεργασία στα πλαίσια της ΚΕΠΑ. Και επίσης, σε στρατιωτικό επίπεδο, το Σεπτέμβριο είχαμε άλλη μια επιτυχία στην ε, συνεργασία, γιατί ένας υψηλά ιστάμενος εκπρόσωπος, ε, από την Ινδονησία ήρθε ε, στην, ε, στις Βρυξέλλες και επίσης πήγε και στην έδρα της επιχείρησης Αταλάντα που είναι μια πολύ σημαντική επιχείρηση και λόγω εντολής αλλά και για την διπλωματία και τη στρατιωτική διπλωματία στη συνεργασία με τους εταίρους ΑΣΕΝ που αυτή τη στιγμή εξελίσσεται πολύ γρήγορα μελλοντικέ προοπτικές που μπορεί να γίνει περισσότερη δουλειά. Τρεις προτεραιότητες βλέπω εγώ. Πρώτον, να ξεπεράσουμε το επίπεδο των σεμιναρίων και διαλόγων και να έχουμε και η επιχειρησιακή συνεργασία. Το μεγάλο ερωτηματικό λοιπόν είναι αυτό, πώς θα το οργανώσουμε. Νομίζω στο μυαλό των ε, Αζεάν πολλές φορές αναρωτιούνται τι μπορεί να προσθέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση πάνω στα σεμινάρια και στο διάλογο. Το είπατε και εσείς, συνεργασία με τα κράτη-μέλη. Τα κράτη-μέλη έχουν στοιχεία ε, στην περιοχή και συνεργάζονται σε στρατητικό επίπεδο καμιά φορά και πολύ μάλιστα. Το ζήτημα είναι πόσο μπορούμε εμείς να παρουσιάσουμε αυτές τις δράσεις υπό το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο μέλλον. Πέραν δηλαδή του στρατιωτικού πεδίου. Γιατί υπάρχουν βαθύτερε εταιρικέ σχέσει, οποίε θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε με του εμπειρογνώμονε των κρατών μελών και των αρμόδιων υπηρεσιών στα πλαίσια τη αντιτρομοκρατία, ε, των υβρεδικών και του κυβερνοχώρου. Δεύτερη ε, πρόκληση συνεργασία και εκτός Ασίας με τους εταίρους μας. Μίλησα για το πλαίσιο και την ετικέτα που είπαμε με και στην Ασία. Δηλαδή, πολύ συχνά μας ρωτάνε τι μπορείτε να κάνουμε παραπάνω εμεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, θα θέλαμε να είναι αφίδρομη η σχέση και ένα συγκεκριμένο τρόπο είναι να προετοιμάσουμε ε, τις αποστολές, ε, του ΟΗΕ, όπου θέλουμε πραγματικά και μα συμφέρει να έχουμε μεγαλύτερη συμμετοχή των Ασιατών σε στρατιωτικό επίπεδο. Θέλουν εκπαίδευση για να το κάνουν και θα μπορούσαμε εκεί εμεί να προσφέρουμε. Και τέλος, να έχουμε καλύτερη επικοινωνία έτσι ώστε να ε, επικοινωνούμε καλύτερα τι επιθυμούμε για το μέλλον. Το αφήγημα, το τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτό το χώρο δεν είναι αρκετά ε, γνωστό. Είναι μια συλλογική προσπάθεια που πρέπει να γίνει και απέτηση και ένα από τα οχήματα τα οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε είναι οι εταιρικές σχέσεις ασφάλειας που θα μπορούσαν με κάποιο απτό τρόπο να ε, ομαδοποιήσουν τις συζητήσεις που γίνονται και βέβαια τις μελλοντικέ συμφωνίε που θα μπορούσαμε να συνάψουμε με τους εταίρους μας, έτσι ώστε να έχουμε μεγαλύτερη ορατότητα. Και το κλείνω εδώ. Sir, now... Σας ευχαριστώ πολύ. Και τώρα η κυρία Πέισοβα. Ε, για το πρόγραμμα της ε, Ασίας, ε, συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω και τον κύριο Εύερτς, λέει η κυρία Πέισοβα, ανώτερη αναλύτρια Ινστιτούτου Μελετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα ασφαλείας. εγώ θα καλύψω ένα κάπως διαφορετικό θέμα και γι' αυτό προσεκλήθη κιόλας, αλλά είναι από τις κρυφές πτυχές ε, των σχέσεων με την Ασία που δεν συζητούμε συχνά. Κανείς σχεδόν δεν το αναφέρει. Και έχει να κάνει με τα όπλα. Πριν φτάσουμε εκεί θα ήθελα να σας δώσω μια επισκόπηση για το πώς έχει αλλάξει το πλαίσιο και το γεωστρατηγικό περιβάλλον που διαμορφώνει αυτή τη στιγμή τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Ασίας. Και μετά θα πάω στην πίεση και στο στην επιρροή της Ένωσης. Μπορεί να έχετε δει πρόσφατα ε, τον όρο Indo-Pacific, Ινδία ε, Ειρηνικός. Έχουμε ξεφύγει από ε, τις Ηνωμένε Πολιτείε και τον Ειρηνικό που είχαν μεγαλύτερο βάρος οι Ηνωμένε Πολιτείε. Και δεν είναι απλώς μια αλλαγή ονοματολογίας αυτή. Είναι μια νέα έννοια που φέρνει την Ασία όλο και πιο κοντά στην Ευρώπη. Ε, μετατοπίζει ολόκληρη την ε, στρατηγική ισορροπία προς δυσμάς, συμπεριλαμβανομένου και του Ινδικού ωκεανού. Αυτό είχε να κάνει με την ασφάλεια στη θάλασσα που ανέφερε προηγουμένως ο Στίβεν και είναι πολύ σημαντικά, αλλά όχι μόνο. Εστιάζει επίσης ε, στα οικονομικά στοιχεία, στο εμπόριο, στη συνδεσιμότητα, όλα αυτά τα καθημερινά λειτουργικά ζητήματα που χρειαζόμαστε. Πώς ξεκίνησε αυτό με την Κίνα και την διαβόητη πρωτοβουλία της ε, ε, μία ζώνη, ένας δρόμος. Ε, το έχουν ονομάσει μάλιστα και το έργο του αιώνα. Το γνωρίζετε η Βαλερή Νικέ, η συνάδελφος από, την, από το ΙΡΙΣ μίλησε για την Αφρική και την Κίνα. Τα γνωρίζετε αυτά τα θέματα. Είναι μια νέα έννοια λοιπόν τώρα και προσπαθούμε να το αντιμετωπίσουμε. Το 2013 ε, ξεκίνησε αυτή η πρωτοβουλία, αλλά το, την τελευταία 20 ετία το εμπόριο διέπει όλη τη διπλωματία της Κίνας. Με τρόπο απλό, ορθολογικό, να κάνουμε επενδύσεις και στατικές υποδομές που βολεύουν στο δρόμο τον εμπορικό. Βέβαια το πρόβλημα είναι ότι υπάρχει και διτή χρήση αυτών των έργων υποδομής ε, λιμένων κτλ. τα έχουμε αναλύσει, δεν θα μπω σε λεπτομέρειες τώρα. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο ανησυχεί την Ευρώπη έτσι άμεσα. Ε, τι έγινε λοιπόν ως απόκριση στην πρωτοβουλία «Μια ζώνη, ένας δρόμος» έχουν αφυπνιστεί οι δημοκρατικές λεγόμενες χώρες ε, ε, σε μία έννοια για έναν ανοιχτό και ελεύθερο ειρηνικό ωκεανό. Από την Ιαπωνία ξεκίνησε αυτό και σε συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες και στρατηγικές μελέτες. Δηλαδή θέλουν να ε, αναζωογονήσουν τις δυνάμεις των ελευθέρων χωρών, των δημοκρατικών χωρών απέναντι στις σκοτεινές επιβολές της Κίνας επιβουλές ε, αναδύεται η Κίνα, ε, αλλά και η Ινδία τώρα ως ε, βασικός πάροχος ασφαλείας στις διμερείς σχέσεις Ιαπωνίας Ινδίας. Αλλά είναι τετραμερής τώρα. Δεν είναι μόνο η Ινδία, η Ιαπωνία και η Αυστραλία που βλέπετε στο χάρτη, αλλά και οι Ηνωμένες Πολιτείες που δεν χωρούσαν στο χάρτη μου. Ε, γίνεται λόγος για κοινέ αρχές και αξίες. Αυτό μπορεί να είναι γενικό και ασαφές. Οτιδήποτε είναι ελεύθερο και δωρεάν ε, και ανοιχτό. Φιλελεύθερες αρχές, ελεύθερη ναυσιπλοεία, κυκλοφορία στη θάλασσα. Ε, κάπως έτσι αρχίζει και διαμορφώνεται αυτή η έννοια και η αντίληψη. Πού καταλήγει. Το περιβάλλον ασφαλείας είναι όλο και πιο βέβαιο ε, ως αποτέλεσμα. Δεν θέλω να σας τρομάξω. Ε, με τίποτα διπολικές αναφορές ε, ψυχροπολεμικού τύπου. Αλλά και εδώ θα μπορούσαμε να διακρίνουμε δύο στρατόπεδα και πρέπει να διακρίνουμε που ε, στατηγικά είναι αντιμέτωπα μεταξύ τους. Πέραν από τις υφιστάμενες εντάσεις που έχουμε με τη Βόρεια Κορέα, την Ανατολική Συνική Θάλασσα, την Νότια Συνική Θάλασσα, την Ταϊβάν κλπ έχουμε και κάποια άλλα υφιστάμενα ε, θέματα που παραγωνίζονται και για την ε, ασφάλεια και την ανασφάλεια. Όταν είναι αβέβαιο το κλίμα, οι χώρες οθούνται στο να θέλουν να λάβουν ε, τα κατάλληλα μέτρα. Δεν ξέρω αν βλέπετε τώρα σε αυτό το χάρτη τις λεπτομέρειες, αλλά αφορούν τις εισαγωγές όπλων των ασιατικών χωρών. Και όπως ίσως γνωρίζετε, η Ασία είναι η Ήπειρος ε, που καταβάλει το μεγαλύτερο ποσό για όπλα, 27%. Ε, ε, μετά τις Ηνωμένε Πολιτείε βέβαια είναι ο μεγαλύτερος εισαγωγέας και είναι λογικό και λίγο κοινικό ότι η ανασφάλεια ευνοεί το εμπόριο και τις business κυρίως για την αμυντική βιομηχανία ε, με μπλε χρώμα εδώ βλέπετε τη συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών στις εξαγωγές όπλων, που είναι ο υπαριθμόν ένα. Με γκρίζο χρώμα είναι η ε, Ρωσία που είναι ο δεύτερος και όλο το κίτρινο είναι ευρωπαϊκές χώρες. Όλη η δυναμική της άμυνας λοιπόν μετατοπίζεται και οι αμυντικές ανάγκες είναι τεράστιες σε βαθμό που έχουν αρχίσει να επενδύουν οι χώρες στην ίδια τους την άμυνα και μετά έχουν αρχίσει να γίνονται ίδιες εξαγωγής όπλων. Αυτό δεν μετατοπίζει απλώς ε, τη δυναμική της παγκόσμιας αμυντικής βιομηχανίας γιατί έχουμε τη Ρωσία και την Κίνα. Καλά, η Ρωσία ανέκαθεν ναι, ήταν εξαγωγές όπλων, αλλά η Κίνα είναι νεοφερμένη και έχουν αρχίσει να είναι και ανταγωνιστικές αυτές προς την ευρωπαϊκή βιομηχανία, ιδιαίτερα η Κορέα, η οποία τώρα εξάγει στο Ηνωμένο Βασίλειο, για παράδειγμα. Θα ήταν όμως αφελές να πούμε ότι το εμπόριο όπλων είναι και αυτό ένα εμπόριο. Όχι, δημιουργεί δεσμούς και εξαρτήσεις. Βλέπουμε χώρες που συνεργάζονται τώρα Κίνα, ε, Ρωσία, ε, η, Κίνα εξάγει στο Μπαγκλαντές, στη Βενεζουέλα, ε, η Ρωσία σε άλλες χώρες και αφρικανικές. Και είναι πολύ ενδιαφέρον να δούμε ότι η Ιαπωνία στρέφεται προς την παραγωγή όπλων τώρα ίδια παρά το διάσημο ειρηνικό και ειρηνιστικό παρελθόν της και το σύνταγμά της. Πώς επηρεάζει τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς μπορεί να έχει σημασία η παρουσία της. Το είδατε από το κίτρινο ε, στην προηγούμενη γραφική παράσταση. Το κλασικό διπλωματικό πακέτο στις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι οικονομικό, πολιτικό, κανονιστικό, όλα αυτά που ανέφερε ο Στίβεν. οικονομική εσοδή, συνεργασία, ε, λειτουργική και επιχειρησιακή κτλ. Αλλά στην ουσία οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν μεγάλο μερίδιο ε, στην αγορά πολλών ε, ασιατικών χωρών. Εξάγουν σε πολλές χώρες. Εδώ ο χάρτης που σας δείχνω είναι λίγο αντιγραφή του προηγούμενου, της προηγούμενης διαφάνειας. Αυτό όμως που μας κάνει ιδιαίτερη εντύπωση και τη μεγαλύτερη, μπορείτε να δείτε εδώ τα ποσοστά ανάλογα με τους υπολογισμούς ποικίλουν. Αλλά σε πολλές χώρες της Νότιο-Ανατολικής Ασίας ε, είναι πάνω από 50% ε, τα όπλα ευρωπαϊκής ε, προέλευσης. 22% του προπολογισμού και παραπάνω. Ιδιαίτερα στη Νότια Συνική Θάλασσα, το έχουμε ξανασυζητήσει, ξέρουμε ότι είναι το υπαριθμόν ένα κρίσιμο σημείο ασφαλείας. Εφτά χώρες συμμετέχουν, έχω βάλει και την Ταϊβάν και το έχω διωγγώσει λίγο, αλλά η Ευρώπη εξάγει όπλα εξίσου και αδιακρίτως προς όλους, συμπεριλαμβανομένης και της Κίνας, που υποτίθεται ότι είναι ο μεγαλύτερος ταραξίας εκεί και υποκινεί τη σύγκρουση. Οπότε αυτό ενέχει το εξής ερώτημα. Εμείς ε, υποδαβλίζουμε αυτή την κούρσα, τον εξοπλισμό. Ποια είναι η στρατηγική θέση και αντίληψη στις Βρυξέλλες ε, ε, απέναντι σε αυτό το τόσο ευαίσθητο θέμα. Και αυτό ήταν και το κεντρικό ερώτημα που ρωτήσαμε σε αυτό το φυλάδιο που σας ε, δείχνω. Σε αυτή τη δημοσίευση του Νοεμβρίου έχω αφήσει στην είσοδο μερικά αντίτυπα. Αυτό είναι το κύριο ερώτημα. Όπως βλέπετε 17% του κινέζικου προπολογισμού ή των εισαγωγών ε, είναι ε, ευρωπαϊκής προέλευσης. Μπορεί κανείς να αναρωτηθεί, μα πώς είναι δυνατόν, αφού έχουμε μπαργκο όπλων. Ε, είναι το, η περίφημη τεχνολογία διτής χρήσης, τεχνολογία και αγαθά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για πολιτικούς και για στρατιωτικούς σκοπούς. Κατά τη διάρκεια των ετών, πολλά τέτοια είδη εξήχθησαν στην Κίνα. Καλά, δεν θα μπω σε λεπτομέρειες. Αεροσκάφη, drones, ε, κινητήρες, χημικά, ε, πυρομαχικά, εκρηκτικά, ε, ραντάρ, σονάρ, ελαφρύς οπλισμός και πάει λέγοντας. Γι' αυτό ονομάζεται και το βιβλιαράκι που βγάλαμε όπλα, κινητήρες και πυρομαχικά. Ε, Πέρα από τα απτά όμως υπάρχουν και μία απτά στοιχεία πολύ πιο δύσκολα να εντοπιστούν. Ε, γιατί πρόκειται για ερευνητική συνεργασία, κοινοπραξίες, ε, σε στρατηγικούς τομείς, συνεργασία κινέζικων με ευρωπαϊκές εταιρείες. Υπάρχει λοιπόν μια δυνατότητα να επηρεάσουμε αν θέλουμε και αν θέλουμε ότι είμαστε σε θέση. Θα ήταν αφελές να πει κάποιος ότι η κούρσα αυτή των εξοπλισμών ή ότι το εμπόριο όπλων είναι και αυτό ένα εμπόριο και όλοι πουλάνε όπλα και παντού στον κόσμο. Ε, αυξάνεται, διευρύνεται το χάσμα μεταξύ της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της πολιτικής των κρατών μελών δημιουργείται μια αμφισημία εδώ. Γιατί αν το δει κανεί ε, ως εξωτερικός παρατηρητής, είναι δύσκολο να πούμε ότι εδώ είμαστε σταθεροποιητικός παράγοντας. Γιατί εμείς ως ερευνητές καμιά φορά ερχόμαστε αντιμέτωποι ε, με ε, έτσι, ακροατήρια που έχουν πολύ μεγάλη ευαισθησία σε αυτά τα θέματα. Έγιναν προσπάθειες συντονισμού, δεν είναι καινούριο αυτό. Η Ευρωπαϊκή Κοινή Θέση του 2008 συνοψίζει τα βασικά κριτήρια ε, συνεργασίας με χώρες, ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων κτλ. Αλλά επειδή δεν είναι δεσμευτικό αυτό και δεν υπάρχει έλεγχος, ε, είναι δύσκολο το θέμα, πόσο μάλλον και τα αγαθάδη της χρήσης. Για να συνοψίσω, Νομίζω ότι αυτά τα θέματα δεν ε, τα αντιμετωπίζουμε. Αυτό που είπε και ο Στίβεν. Αλλά για να πω και κάτι θετικό κλείνοντας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρείται σημαντικότερος παράγων ασφαλείας ακριβώς λόγω ε, του ρευστού γεωστρατηγικού περιβάλλοντος. Για να το πω, μα δεν μπορούμε πλέον να ε, υπολογίζουμε στις Ηνωμένε Πολιτείε ως βασικό πάροχο ασφαλείας. Η Ιαπωνία, η Ινδία, η Αυστραλία προσβλέπουν και θα καλωσόριζαν μια ε, πιο ε, έντονη ευρωπαϊκή ε, παρουσία. Και η ΠΕΣΚΟ και οι άλλες πρωτοβουλίε που έχουμε, η μόνιμη διαρθρωμένη συνεργασία, είναι πρόσδεκτα. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση μετακινείται από το παλιό καθεστώς της πολιτικής δύναμης με, τον, τη μη στρατιωτική έννοια του όρου δηλαδή. Και ακριβώς αυτό το θέμα θα πρέπει να μας απασχολήσει και να το εξετάσουμε. Σταματώ εδώ. Ευχαριστώ. I would like to thank... Ευχαριστώ και τους δύο μιλητές. Πολύ ενδιαφέρουσες οι παρουσιάσεις τους, ε, λίγο ανησυχητικές. ενθαρρύνω του βουλευτέ που είναι παρόντε να πάρουν το λόγο. Ο κύριο Πάσκου θέλει να πάρει το λόγο. Κατανάγκη. Κατά ανάγκη. Γιατί ο άλλος συνάδελφο από το ΕΛΚ δεν είναι εδώ. Είναι η κυρία Σουίτσα βέβαια, Σουίσα. Άκουσα μόνο το τέλος παρουσίασή σας, κυρία μου. Και αυτά είναι δεδομένα που δεν θα περιμέναμε να ακούσουμε. Πάντως όποιος διαβάζει ανακαλύπτει. Και αν τα διαβάσει, κανεί, κανείς θα τα ανακαλύψει αυτά. Η Έμα, η Εύα, είπε ότι η γεωπολιτική της περιοχής έχει αλλάξει. Και έχει αλλάξει και η ελκυστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για άλλα κέντρα εξουσιών. Συμφωνώ, είναι αλήθεια αυτό. Επομένως, ρωτώ το εξής. Υπάρχει ένας παγκόσμιος ανταγωνισμός ανάμεσα στις δύο υπερδυνάμεις την, ε, της ΙΠΑ και την Κίνα. Εμείς έχουμε συμφέροντα. Συμπίπτουν απόλυτα τα συμφέροντά μας με των ε, Αμερικανών. Γιατί καταλαβαίνω τους Αμερικανούς και προσπαθώ να καταλάβω και τους Κινέζους, αλλά τους Αμερικανούς καταλαβαίνω θέλουν να επιβραδύνουν λιγάκι και αν μπορούν να εξαλείψουν την, τον ανταγωνισμό της Κίνας και να μην φτάσει στο επίπεδο να γίνει πραγματική υπερδύναμη η Κίνα. Ωραία, καλά και άγια όλα αυτά, αλλά εμείς που βρισκόμαστε είναι μενόμενο να συνταχθούμε 100% με τους Αμερικανούς. Έχουμε δικά μας συμφέροντα απέναντι στην Κίνα. Σε ποιο βαθμό είναι ανταγωνισμός απέναντι στην Κίνα αυτή η σχέση και σε ποιο βαθμό είναι συνεργασία, όχι μόνο στο στρατιωτικό τομέα, αλλά και επέκεινα. Χρειαζόμαστε μία ανάλυση με περισσότερες αποχρώσεις, περισσότερες λεπτομέρειες, ποια είναι η θέση μας σε αυτή τη νέα αντιπαλότητα που υπάρχει ανάμεσα στις υπερδυνάμεις. Η κυρία Λόιζινγκ. Ευχαριστώ πολύ. Θα μιλήσω γερμανικά. Περιμένω να βάλετε τα ακουστικά σας. Πρώτη ερώτηση προς την κυρία Πέσοβα ειδικά. Εσείς ζητάτε πιο ενισχυμένο ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι ε, απλώς μεμονωμένων κρατών μελών στον ειρηνικό. Δύο ερωτήσεις έχω εγώ. Τι εννοείτε και στρατιωτική παρουσία ε, ως αποστολή ΕΠΑΑ ή κάποια διαφορετική παρουσία. Και αν ναι, τι ακριβώς έχετε στο μυαλό σας. Δεύτερη ερώτηση. Θα πρέπει να επεκταθώ. Στις 11 Φεβρουαρίου ξαφνικά ο Γκέβιν Βίλιαμσον, ε, υπουργό Αμήνη του μενού Βασιλείου, ε, έκανε μια ομιλία θέσεων ε, για την διεύρυνση της στρατιωτικής παρουσίας στον Ειρηνικό. Αυτό τον καιρό τέτοιες πρωτοβουλίες ε, φαίνεται να ε, είναι κάτι το διμερές, ε, Ηνωμένο Βασίλειο Γαλλία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι τελείως απ' έξω, γιατί από ό,τι φαίνεται δεν είναι επιθυμητή μια εμπλοκή της. Στην εφημερίδα Frankfurt Allgemeine πρόσφατα, που είναι μια πολύ συντηρητική γερμανική εφημερίδα, δημοσιεύθηκε ένα άρθρο ε, που ε, θεωρεί αυτές τις γαλλοβρετανικές προσπάθειες ως απειλή για τα γερμανικά συμφέροντα. Και παραθέτω, θέλουν να διευρύνουν ε, Βρετανία και Γαλλία τη στρατιωτική τους επιρροή στην Άπο Ανατολή. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να υποστηριχθούν από τη Γερμανία για να έχουν οι Βρετανοί εμπορικά πλεονεκτήματα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. και ε, κινδυνεύει να ε, υπάρξει και σύγκρουση Γαλλίας-Γερμανίας. Γιατί αυτό που ενδιαφέρει τη Γαλλία είναι να έχει κέρδη η δική της αμυντική βιομηχανία και να αποκλειστούν άλλοι ανταγωνιστές όπως είναι η γερμανική ε, βιομηχανία. Υπογραφή Björn Müller, που είναι ξέχων στέλεχος της γερμανικής έτσι, στρατηγικής ελίτ. Εσείς πώς τα αξιολογείτε όλα αυτά, η κυρία Αναγκόμες. Μικρόφωνο παρακαλούμε για την κυρία Γκόμες. The shocking Σοκαριστικό το συμπέρασμα και σας ευχαριστώ ε, για το γεγονός ότι μας διαβιβάσατε αυτά τα μηνύματα. Αυτό τι δείχνει, δεν υπάρχει Ευρώπη. Όταν υπάρχει Ευρώπη, παραβιάζει τους δικούς, τους, τους δικούς τους κανόνες. Έχουμε κοινή θέση για την εξαγωγή όπλων. Και προσπάθησα ε, το 2009 να κάνω πολύ, έκανα πολλή προσπάθεια για να καταστεί δεσμευτική αυτή η θέση. Και παραβιάζεται. Αυτό είναι η απόδειξη λοιπόν ότι δεν υπάρχει Ευρώπη. Και ακριβώς γι' αυτό το ερώτημά σας για την στρατηγική, το στρατηγικό προβληματισμό ποιο είναι. Λεφτά στις πρωτεύουσε. Στις, ε, στις τώρα ο στρατηγικός προβληματισμός, ε, η στρατηγική σκέψη και αν υπάρχει, δεν ενδιαφέρεται κανένα. Αμφισβητείται λοιπόν η Ευρώπη και τα συμφέροντα για την ασφάλεια της Ευρώπης αμφισβητούνται από τα κράτη-μέλη. Και το λέω, μα, περί αυτού πρόκειται. Το δικό μου ερώτημα τώρα ποιο είναι. Για τις εξαγωγές ε, αγαθών διπλής χρήσης. Ε, είναι πολύ πιο σοβαρό από τα συμβατικά όπλα. Φυσικά τα συμβατικά όπλα ε, έχουν τεράστια επίπτωση στις κοινωνίες και στον έλεγχο των κοινωνιών. Φυσικά η Ευρώπη φταίει, τα κράτη-μέλη φταίνε για το γεγονός ότι στην πραγματικότητα κάλεσαν την Κίνα να έρθει και να αγοράσει φθηνά τις αμυντικές μας, βιομηχανίες, ε, και στη χώρα μου και παντού ξεπουλήσαμε στην Κίνα τι αμυντικέ μας βιομηχανίες. Και δεν μίλησατε καθόλου για τα πυρηνικά. Όταν μιλάμε για αυτή την αντιπαλότητα για την οποία μιλήσατε και βάλουμε μέσα στην εξίσωση και τα πυρηνικά, το πράγμα γίνεται πολύ πιο σοβαρό για την ανθρωπότητα, αλλά και ιδίως για την Ευρώπη. Δεδομένου ότι υπάρχει και το Πακιστάν που έχει πυρηνικά και η Ινδία εκτός της συνθήκης. Το Πακιστάν. Ε, οι, Σαουδάραβες έχουν πακιστανικά όπλα. Δεν το έλεγαν ότι τα είχαν αγοράσει από, την, από το Πακιστάν. Όταν βλέπουμε τι γίνεται επίσης με τη συνθήκη για τα πυρηνικά μεσαίου βεληνικούς, πρέπει να δούμε το ρόλο της Κίνας. Τι θα γίνει με το νέο start και τα λοιπά. Θα μπορούσατε να μιλήσετε λίγα και αυτά τα θέματα. Ευχαριστώ. Να θέσω κι εγώ ερωτήματα. Ε, και στους δύο, αλλά κυρίως στην Εύα Πέσοβα. για την συνεργασία για θέματα ασφάλειας και την αντιπαλότητα που υπάρχει μεταξύ Κίνας και Ρωσίας. Μιλάμε για την ασφάλεια και την άμυνα. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Στίβεν Έβερτς πρώτα και μετά στην Εύα Πέσοβα. E <laughs> Σύμβουλος στην ΕΙΑΔ και μετά στην ε, Εύα Πέσοβα. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να απαντήσω. Είναι κανένα δύο ερωτήσεις που συνδυάζονται περισσότερο με τα όσα είπα εγώ και κάποια που θα έπρεπε να απαντήσει η Εύα. Να σας πω πως Πραγματικά θα έπρεπε να σας ε, ε, χειροκροτήσουμε για το γεγονός ότι θέσατε το θέμα αυτό στο τραπέζι. Γιατί είναι ζήτημα βέβαια που κυρίως θα πρέπει να σκεφτούν τα κράτη-μέλη για το τι δηλαδή επιθυμούν ε, και ποιες θα είναι οι συνέπειες. Δεν είναι προφανή ε, τα συμπεράσματα μπορούν να ακολουθήσουν διαφορετική κατεύθυνση και δεν υπάρχει μόνο ένα μήνυμα ε, το οποίο παίζει εδώ. Είναι πολλά τα μηνύματα και χρειάζονται μια σε βάθο συζήτηση η οποία ακόμα δεν έχει γίνει. Για την ευρύτερη γεωστρατηγική ερώτηση του πού τοποθετεί ε, τον εαυτό της η Ευρώπη στην ε, ε, εντατικοποιημένη μάχη για την πρωτοκαθεδρία, να σας πω πως σε πολλούς χώρους αυτό το οποίο έχουμε αποκρισταλώσει και αυτή είναι η μεγαλύτερη τάση στις παγκόσμιες, στην παγκόσμια σκηνή και κυρίως στην πολιτική παρουσία της Κίνας και της Ασίας, το θέμα είναι το εξής. Εμείς θα πρέπει να υπερασπιστούμε τα ευρωπαϊκά συμφέροντα και όχι να το προσεγγίζουμε ε, μέσω αυτής της ε, ε, μονοδιάστατης προσέγγισης στο με ποιον είσαι. Όχι, είμαστε με την Ευρώπη, με τα ευρωπαϊκά συμφέροντα. Και θέλουμε να στηρίξουμε την σταθερότητα, την ειρήνη το να είμαστε ανοιχτοί στην, στην ευρύτερη περιοχή ε, ε, της Ασίας και του Ειρηνικού. Δεν είναι μια διπολική ερώτηση, δεν είμαστε με τον ένα ή με τον άλλον. Πολλοί έχουν αυτή την ε, προσέγγιση και βέβαια στην πολιτική πολλές φορές πρέπει να κάνεις μια επιλογή. Αλλά για την ασιατική πολιτική νομίζω η ορθότερη λύση είναι ακριβώς το να μην διαλέγεις ε, κάποια πλευρά. Δεν είναι αυτό μια παρελκυστική τακτική, δεν είναι έλλειψη επιλογών, όχι. Ε, νομίζω ότι ε, για τη ΣΥΠΑ αυτό είναι πολύ προφανές ότι ακολουθούν μια πολύ πιο σκληρή προσέγγιση με την Κίνα ε, ενώ εμείς ακολουθούμε μία τριπλή προσέγγιση. Έχουμε σημεία στα οποία, και κεφάλαια με τα οποία συνεργαζόμαστε εξαιρετικά με την Κίνα και είναι πολύ σημαντικά για μας, αλλαγή του κλίματος και άλλες διεθνείς συμφωνίες. Κάποιους χώρους με τους οποίους χρειάζεται να διαπραγματευτούμε πολύ σκληρά μαζί τους επενδύσεις, αμοιβαιότητα. Και επίσης υπάρχουν και θέματα στα οποία είμαστε στρατηγικοί ανταγωνιστές με την Κίνα. Και αυτό θα πρέπει να το έχουμε ξεκάθαρο. Όμως επαναλαμβάνουν αυτή η τριπλή ε, προσέγγιση και στις ΙΠΑ νομίζω ακολουθούν μία μονοδιάστατη ε, προσέγγιση και τα βάζουν όλα στο ίδιο καλάθι, κάτι το οποίο για μας δεν είναι η σωστή προσέγγιση. Και μέσα σε αυτό το ευρύτερο πλαίσιο να πω δύο λέξεις για την Κίνα και τη Ρωσία. Η δική μου γραμμή είναι ότι εμείς δεν έχουμε κανένα συμφέρον στο να τους φέρουμε πιο κοντά από τη στιγμή που δεν βρίσκονται τόσο κοντά. Πολλές φορές δίνουμε την... Ε, υπάρχει εντύπωση που υπάρχει νέα γεωστρατηγική συμμαχία μεταξύ Πεκίνου και Μόσχας και πολλές φορές λόγω τακτικών επιλογών, επιλογών τακτικής αυτό συμβαίνει, δεν ε, το αποκλείω, το βλέπω. Αλλά γενικότερα εμείς έχουμε γεωστρατηγικά συμφέροντα. Μας είπατε γεωστρατηγική σκέψη. Ο γεωστρατηγικός στόχος είναι να μην ενισχύσουμε εμείς την συμφωνία και τη συμμαχία μεταξύ Ρωσίας και Κίνας γιατί δεν είναι τόσο ισχυρή αυτή τη στιγμή όσο κάποιοι φαντάζονται. Λοιπόν, και για την Κίνα και για το θέμα Ρωσίας Κίνας, να μην μπούμε εμείς στα στεγανά και φυλακιστούμε μέσα σε αυτή την συνεργασία και σημασία μεταξύ τους, την οποία εμείς θα χτίσουμε. Είπαμε, Αζεάν, Αυστραλία, Ινδία είναι πολλοί παίκτες που όπως και εμείς δεν θέλουν να σκληρύνουν ε, τις θέσεις ε, και τα στρατόπεδα. Η κυρία Πέσοβα. Θα συμφωνούσα πως θα ήταν κάπως απλουστευτικό και δεν θα πρέπει να το δούμε ως ε, διπολικό, διπολική επιλογή μεταξύ Κίνας και είπα, υπάρχει κάποιο είδος διπολισμού και έχει να κάνει με τις αξίες που εκπροσωπούν, αλλά ναι, αν θέλουμε το κράτος δικαίου, ναι, ε, έχουμε τον κίνδυνο αναρχίας που ε, βρίσκεται μέσα σε αυτή την μερκαλιστική, μερκαντιλιστική άναρχη και άγρια πολιτική που ακολουθεί η Κίνα. Ναι, αλλά και στη στρατόπεδο των ΗΠΑ υπάρχουν και πολλέ χώρε που έχουν τα δικά του συμφέροντα. Οπότε αυτό που αντιμετωπίζουμε είναι έναν πολυκεντρικό πλανήτη όπου όλοι οι παίκτε υπερασπίζονται τη δική του γειτονιά, τα δικά του συμφέροντα και τα δικά μα συμφέροντα είναι κράτο δικαίου. Και νομίζω ότι το μέτωπο είναι ευρύτερο από αυτό που κάποιοι πιστεύουν. Πρέπει να βρούμε απλώ τα κατάλληλα εργαλεία. Θα συμφωνήσω για το θέμα Ρωσίας-Κίνας. Εμείς μεγενθύνουμε αυτή την σχέση. Γιατί και πάλι μοιάζει να είναι προφανής, γιατί είναι στην άλλη πλευρά αυτού του σχεδίου αξιών που μόλις περιέγραψα, του συστήματος αξιών, αλλά αν τις δείτε από κοντά είναι ανταγωνιστές και δεν συμπαθούν η μία την άλλη. Συνεργάζονται μεν ε, με έναν ελάχιστο κοινό παράγοντα και στα πλαίσια της διάσκεψης Σανγκάης, αλλά είναι ανταγωνιστικές χώρες στην Κεντρική Ασία, για παράδειγμα, που είναι η γειτονιά τους. Και έχουν βασικές διαφορές εκεί, οπότε σας παροτρύνω να ε, διαβάσετε μία ακόμα δημοσίευση των συναδέλφων μου, κυρία Πρόεδρε, ακριβώς για το θέμα αυτό, για την στρατιωτική βιομηχανία της Κίνας και της Ρωσίας και οι δύο είναι τεράστιες βιομηχανίες. Κυρία Λέοζεν, τι είδους στρατιωτικές αποστολές θα μπορούσαμε να προβλέψουμε για την Ευρώπη στην περιοχή αυτή. Μία που ακούγεται όλο και πιο συχνά είναι η θαλάσσια ασφάλεια. Γενικότερα, που θα βασίζεται στις υφιστάμενες προσπάθειες που γνωρίζουμε, η επιχείρηση Αταλάντα, υπάρχει ο πολιτικός μηχανισμός που μας επιτρέπει να δημιουργήσουμε ένα στόλο και βεβαίως να επεκτείνουμε αυτή την αποστολή και την εντολή της. Δεν λέω την Αταλάντα συγκεκριμένα, αλλά υποθετικά ομιλώντας, εάν πρόκειται να μιλάμε για στρατιωτική αποστολή, θα μπορούσε να είναι συμβολική ε, μασία στην άμυνα τη ελευθερία πλοήγηση. Και όχι απαραίτητα όπω κάνουν οι Αμερικάνοι, αλλά πιο πολύ ευθυγραμμισμένοι με το όσο κάνουν οι Γάλλοι. Και αυτό έχει ήδη συμβεί στα πλαίσια της αποστολής Jean d'Arc πριν από δύο χρόνια, όπου είχαμε ευρωπαϊκή παρουσία επαρκή, γιατί ουσιαστικά είναι ο συμβολισμός της παρουσίας και αυτό για τις χώρες ΑΣΕΑΝ ήταν αρκετός για να αναγνωρίζουν πως η Ευρώπη έχει συμφέρον στην ε, περιοχή και ε, πρόκειται να τα υποστηρίξει. Έχουμε και άλλε χρήσει, δεν τι έλεγα στρατιωτικέ αποστολέ, γιατί δεν είναι πάντα στρατιωτική η στόχη μα. Δεν υπάρχει αυτή η ανάγκη. Υπάρχουν τόσοι πολλοί στρατιωτικοί παίκτε στην περιοχή. Η δική μα δύναμη είναι το ότι είμαστε διαφορετικοί και ακριβώ στηρίζουμε το κράτο δικαίου και εστιάζουμε στα πρακτικά ζητήματα της συνεργασίας, για παράδειγμα, ε, ε, πληροφορίες, ενημέρωση, αλληλεπικοινωνία κτλ. Για την παρουσία του Ηνωμένου Βασιλείου, αυτό δημιούργησε πάρα πολλές αντιδράσεις οι συνάδελφοι που παρακολουθούν τα θέματα θαλάσσιας ασφάλειας στην περιοχή εκεί θεώρησαν πως ήταν αρκετά διασκεδαστική αυτή η ιδέα γιατί το Ηνωμένο Βασίλειο ήδη βρίσκεται στην περιοχή. Πάρα πολύ. Πάντα ήταν. Είναι ε, μία από τις πέντε δυνάμεις με τη Σιγκαπούρη, Αυστραλία, Μαλαισία και ΗΠΑ. Ε, κάνει γυμνάσια πολύ συχνά στην περιοχή. Έχει βάση το Μπρουνάι. Έχει σταθμό στη Σιγκαπούρη. Δεν χρειάζεται δηλαδή να, ενθα... να ενδυναμώσει την παρουσία του, οπότε από πλευρά Υπουργό Άμυνα θεωρώ πω ήταν μάλλον μια ρητορική ε, έκφραση για να δείξει την αποφασιστικότητα τη χώρα να επιστρέψει στην περιοχή. Αλλά δεν χρειάζεται να επιστρέψει, είναι ήδη εκεί. Και πολύ μάλιστα. Οπότε να σας πω ότι υπάρχουν και άλλα που είναι εκεί και δεν θα έπρεπε αυτό να αποτελεί πρόβλημα. Η Γαλλία είναι εξαιρετικά παρούσα η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να χρησιμοποιήσει θετικά αυτή την παρουσία, γιατί αν θέλει κανείς να πει έχουμε συμφέρον, μπορείτε έχουμε συμφέρον και κοιτάξτε τι κάνουν οι Γάλλοι για παράδειγμα. Και αν δει κανείς την, Ινδο, την στρατηγική της Γαλλίας για την Ανδία και τον Ειρηνικό, ευθυγραμμίζεται με τις αρχές της ευρωπαϊκές. Οπότε νομίζω ότι μπορούμε να έχουμε αμοιβαία στήριξη και αυτό είναι το θετικό. Κυρία Γκόμες. Πυρηνικά, απόσυρση από τη σχετική συμφωνία, όντως είναι μεγάλο πρόβλημα που θα το συνέδεια με, την... με τα όσα είπα στην αρχή των απαντήσεών μου. Δηλαδή, τέτοιου είδους εξελίξεις, δηλαδή η ΕΠΑ και το γεγονός ότι αποσύρονται από τη συμφωνία αυτή, υποσκάπτουν τη θέση των ΕΠΑ σε κάποιο βαθμό και δημιουργούν την ανάγκη να μπουν άλλοι παίκτε. Και αυτό θα μπορούσε να είναι και η Ευρώπη που θα επιστρέψει στο προσκήνιο. Και αυτό το καταλαβαίνουν πολύ καλά οι μεγάλοι παίκτε στην περιφέρεια. Ξέρουμε πως έχουμε ε, κάποιες ε, θέσεις default, αλλά κράτος δικαίου, ε, μη διάδοση πυρηνικών, όλα αυτά τα θέματα τα έχουμε ε, εκφράσει πάρα πολύ στεναρά και ακριβώ επειδή είχαμε τέτοιου είδου αποσύρσει από τη συμφωνία, θα μπορούσε η Ευρωπαϊκή Ένωση να ε, ε, δυναμώσει τη φωνή της, αλλά θα πρέπει να αναλάβουμε και την ευθύνη των πράξεών μας. Wow. I think... Λοιπόν, νομίζω ότι ο χρόνο μας, σχεδόν έχει τελειώσει. Ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους εξαιρετικούς ομιλητές μας, την Συμπρόεδρο, την Μπραφ Σουίτσα, για την διεύθυνση τη συζήτηση για τα δύο αυτά θέματα που είχαμε σε κοινή συνεδρίαση με την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Παρακαλώ να παραμείνετε. Έχουμε και άλλο θέμα ε, το πρωινό, αφού αλλάξουν τα μέλη του Προεδρείου. Ανταλλαγή απόψεων με τον στρατηγό Κλάοντιο Γκρατσιάνο, πρόεδρο της Στρατιωτικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Σε λίγα λεπτά θα αρχίσει η συζήτηση αυτή. Ας χειροκροτήσουμε λοιπόν από κοινού τους ομιλητές μας. Thank you once more.